που έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, όπως ισχύουν και για τα προϊόντα που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τις επεξηγήσει ψήφου. Τα πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο σώμα στην αρχή τη επόμενης ε, συνόδου. Τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν θα πάνε στους, ε, στον προορισμό τους. Εδώ διακόπτεται η περίοδο συνόδου και τελειώνει η συνεδρίασή μας. <laughs>